Έχουν πάρθει φωτογραφίες, τώρα μπορείτε να καθίσετε. Ε, μετά από ακρόαση του κυρίου Κόρβιν Μίχια και βάσει του άρθρου 166 του κανονισμού του Κοινοβουλίου, αποφάσισα να επιβάλλω στον βουλευτή αυτό μία κύρωση για τις απαράδεκτες του παρατηρήσεις για τους Αφρικανούς μετανάστες στην ε, Ολομέλεια της 7ης Ιουνίου. Θα εφαρμοστεί λοιπόν μία πίνη στον κύριο Κόρβιν Μίχια ο κύριος και χάνει το δικαίωμά του σε per diem για μια περίοδο 10 ημερών και επίσης αναστέλλεται η συμμετοχή του σε όλα τα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 5 συνεχείς ημέρες. Από τις 12 Σεπτεμβρίου ξεκινά η εφαρμογή αυτής της ποινή προς τον κύριο Κόρβιν Μίχη. Η απόφαση αυτή έχει κοινοποιηθεί χθες στον κύριο Κόρβιν Μίχη. Και θα ήθελα να αναφέρω να πω ότι ο κύριος Κόρβιν Μίκε έκανε και πάλι στην πρόσφατη Ολομέλεια δηλώσεις οι οποίες θα ελεγχθούν κατά πόσο έχουν ρατσιστικό χαρακτήρα και μπορεί να επισύρουν περαιτέρω κυρώσεις εναντίον του. Ερχόμαστε στη διαδικασία ψηφοφοριών. η κατάσταση των ανθρώπων με αλφισμό στην Αφρική και ιδίως στο Μαλάουι. Ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία.